Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Έχετε φέρει όλοι τις κάρτες ε, για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Περνάμε στο πρώτο σημείο, την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Χιλής για το εμπόριο βιολογικών προϊόντων. Όπως ξέρετε, η συγκεκριά μας είναι η κυρία Κριστίνα Αγγιλέρα και αρμόδια καθήλων επιτροπή, Επιτροπή Εσωτερικού, Εσωτερικής Αγοράς. Καλύτερα να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, τη συντάκτηρα γνωμοδότησης, για να μας ενημερώσει. Αν το επιθυμεί φυσικά, η κυρία Αγγιλέρα. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας καταρχήν. Όλοι γνωρίζετε ότι η μοναδική δυνατότητα που έχουμε εμείς η Επιτροπή, ως Επιτροπή είναι να πούμε ναι ή όχι, να δεχτούμε ή να απορρίψουμε την πρόταση. Γνωρίζω ότι επιλήθηκε του θέματος ο πρόεδρος μας, αλλά στις συνθήκες όταν ε, όταν αναφέρονται σε ζητήματα για γεωργικών προϊόντων και διατροφής, ε, αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή πρέπει να είμαστε εμείς, όχι Επιτροπή ε, διεθνού Εμπορίου. Σε τέτοια όμως είναι κρίμα που σε τόσο σημαντική εμπορική συμφωνία μπορούμε απλώς να πούμε ναι ή όχι, να δεχτούμε ή να απορρίψουμε τη συμφωνία. Και αυτό επιδιώκει ο πρόεδρος μας τώρα με τα διαβήματά του, στο μέλλον να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση τέτοιων συμφωνιών. Προς το παρόν όμως, επαναλαμβάνω, μόνο αποδοχή ή απόρριψη μπορούμε να, κρατήσουμε μόνο αυτή τη θέση, να υιοθετήσουμε. Εγώ προτείνω αποδοχή της συμφωνίας. Άλλωστε, ε, τώρα πρόκειται να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα εγώ το αναφέρω σε αιτιολογική σκέψη αυτό, γιατί η θέμα μα είναι να δεχτούμε ή να απορρίψουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δική μου σύσταση, η δική μου πρόταση στη γραμμοδότηση είναι να εγκρίνουμε τη συμφωνία, αλλά στο μέλλον να διεκδικήσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή τη Επιτροπή Γεωργία, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι σήμερα, που περιορίζεται σε ναι ή όχι. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε. Στη διάσκεψη, στη διάσκεψη Προέδρων είχα την ευκαιρία να αναπτύξω το θέμα πιο διεξοδικά όταν σας αντικατέστησα και ελπίζω στο μέλλον να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και να ακούγεται περισσότερο ο λόγος μας σε τέτοιου είδους συμφωνίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Αγγιλέρα. Αναφέρθηκε το ζήτημα στη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά θα επαναλάβουμε το εγχείρημά μας το διάβημά μας και γραπτός, διεκδικώντας κάποιες διορθώσεις, όχι μόνο σε θέματα κατανομής αρμοδιοτήτων, αλλά και διαδικασίας. Θα αναλάβει η Γραμματεία την εκπόνηση της πρότασης που θα υποβάλει προς έγκριση στους συντονιστές. Μετά τις παρατηρήσεις κυρίας Αγγιλέρα της συντάκτηρης γνωμοδότης, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε δύο τροπολογίες μόνο που είναι και πανομοιότυπες, θα τις ψηφίσουμε διανατάσσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ των δύο τροπολογιών, ένα και δύο υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Οπότε ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Οπότε τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση της κυρίας Αγγιλέρα. Συγχαίρομαι τη συντάκτριά μας. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες. Ο κύριος Ντές έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για την προστασία των εργαζομένων και μετά από τις πρόσφατες ε, καταστροφές στην Πορτογαλία. Oh. Gerade als sollten wir Opfer gedenken. Νομίζω ότι πρέπει καταρχάς ε, να αφιερώσουμε ένα λεπτό για να τιμήσουμε τα θύματα της καταστροφής. Ε, Πολύ καλή πρόταση. Θα τηρήσουμε ένα λεπτού σιγή. Bardzo dziękuję. Και επανερχόμαστε στο σημείο 7, την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους ε, συναφείς με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Η συγκεκριτή μα συντάκτης είναι ο κύριος Ζωζέ Μποβέ, ενώ αρμόδια καθήλυνα επιτροπή είναι η Επιτροπή Απασχόλησης. Φυσικά οι απασχολούμενοι στον αγροτροφημικό κλάδο εκτίθενται σε μια σειρά από ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες ή να οδηγήσουν σε διαταραχές και καρκινο, καρκινογόνα αποτελέσματα. Οπότε θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέτρα για να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στην ε, Ήπεθρο και σε γεωρικές δραστηριότητες. Στις 21 Μαρτίου αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση επί της νομοθετικής πρότασης ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Την γνωμοδότηση την ανέλαβαν οι πράσινοι και όρισαν συντάκτη της γνωμοδότησης τον κύριο Μποβέ. Στον εισηγητή μας θα δώσω το λόγο για να μας κάνει την εισαγωγή. Κύριε Μποβέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια γνωμοδότηση για πέντε προϊόντα. Δεν μιλάμε για όλα τα χημικά προϊόντα. Είναι οκτώ ε, προϊόντα ε, ορυκτά ελαία. Ορυκτά που είναι μεταλλαξιογόνα. Η γνωμοδότηση είναι σωστή. Η έκθεση πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Νομίζω όμως... Δεν με ακούτε. Έχουμε πρόβλημα με τη γαλλική διερμηνία. Już może będzie dobrze. Bardzo proszę, panie pośle, proszę kontynuować. Είναι μια γνωμοδότηση που αφορά πέντε ειδικά προϊόντα που είναι ορυκτέλεια και μηχανέλεια. Μιλάμε ε, για προϊόντα που εντάσσονται σε ένα πολύ πιο ευρύ σύστημα. Είναι όμως η, η δική μας μια πολύ συγκεκριμένη ε, γνωμοδότηση για αυτά τα προϊόντα. Από αυτή λοιπόν την έκθεση μπορούμε και ακριβώς γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε εμεί που ασχολούμαστε με τα γεωργικά, να πάμε πιο μακριά, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την προσπάθεια της Κομισιόν. Τέτοια, τέσσερα σημεία πολύ συγκεκριμένα. Σήμερα ο καρκίνος είναι ο πρώτος ε, λόγος θανάτου ε, στο χώρο εργασία, 53% ε, των θανάτων προκαλούνται από καρκίνο. Θα πρέπει λοιπόν η νομοθεσία να είναι πιο προστατευτική αυτό είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης και εμείς προτείνουμε στη γνωμοδότησή μα να πάρουμε ως αναφορά το, τη χαμηλότερη τιμή με βάση το τι ισχύει στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μοιράσατε σε όλους τον κατάλογο των 28 ε, χωρών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα μέτρα που προωθεί κάθε κράτος για αυτά τα προϊόντα και κατά την το κείμενό μας, συστηματικά βάζουμε ως πρόταση τη χαμηλότερη τιμή που υπάρχει σε οποιοδήποτε κρατό μέλος για να προστατεύσουμε καλύτερα τους εργαζόμενους. Τρίτον, προσθέσαμε σε αυτή την κνομοδότηση γιατί δεν υπήρχε στην πρόταση της ε, Κομισιόν, τους γεωργούς, οι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη γιατί μιλάμε γενικά για εργαζόμενου. Στην πραγματικότητα όμω οι γεωργοί, οι αγρότες δεν προστατεύονται σημαντικά. Είναι σημαντικό για μας να προστατεύονται και οι αγρότες, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι μισθωτοί. Τέλος. Στην γνωμοδότηση αυτή τονίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε καλή προσπάθεια γιατί ενσωμάτωσε το σύνολο των επιστημονικών θέσεων, των ε, διεθνών επιτροπών, παραδείγματος χάρη της ε, ΠΟΗ και τα λοιπά, στην προσπάθειά της. Είναι σημαντικό λοιπόν να τονιστεί αυτό. Αυτό το κείμενο πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Ε, θέλαμε απλώς να διορθώσουμε κάποια στοιχεία του κειμένου της Κομισιόν για να είναι ακόμα καλύτερο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Περνάμε στη συζήτηση. Το λόγο έχει ζητήσει πρώτα ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή και συμφωνώ ανεπιφύλακτα με την πρόταση να επεκτείνουμε την κατηγορία των αναγκαζομένων που καλύπτονται από την οδηγία σε όλους τους εργαζόμενους στη Γεωργία. Γιατί καθημερινά έχουμε έρευνες που αποδεικνύουν ε, την συνάφεια της έκθεσης ε, ε, σε τέτοιες ουσίες και της ανάπτυξης εμφάνισης ασθενειών. Οπότε είναι σημαντικό να εντείνουμε την προστασία. Επίσης θέλουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά την κατηγορία των εργαζομένων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. μου θα ήταν μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα και το γνωρίζουμε, ε, το είδαμε και επ' ευκαιρία τη συζήτηση για την γλυφοζάτη, ε, θα πρέπει να μας δώσει ένα κατάλογο κριτηρίων και τη διαδικασία που ακολουθεί για να ε, εντάξει τις χημικές ουσίες στις καρκινογόνες. Πρέπει να αποφύγουμε τους κινδύνους από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Επίσης, θέλουμε ιδιαίτερη προσέγγιση ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και πώς ε, καταλήγουμε στο χαρακτηρισμό μιας ουσίας ως καρκινογόνου. Γιατί είναι επίμαχο το θέμα του κατά πόσο η γλυφοσάτη είναι καρκινογόνος ουσία. Γιατί δίστανται οι ακόμη και μεταξύ των επιστημόνων. Δεν υπάρχει μια ομοιόμορφη επιστημονική άποψη και γι' αυτό είναι δύσκολο και για μας τους νομοθέτες να αποφασίσουμε ποιος είναι ο κίνδυνος και ο αντίκτυπος για την ανθρώπινη υγεία, αν ούτε οι επιστήμονες δεν συμφωνούν. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερη συνοχή, συνα, συνάφεια στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περισσότερη διαφάνεια για θέματα που είναι όλο και πιο ευαίσθητα για την κοινή γνώμη, γιατί και η κοινωνία ευαισθητοποιείται για τα θέματα αυτά. Και αν θέλουμε να αναπτύξουμε τους δεσμούς και τη σχέση των γεωργών με τους καταναλωτές, φυσικά έχουμε καθήκον να να χειριστούμε το θέμα όπως το κάνει ο Ζωζέ στην γνωμοδότησή του, δηλαδή με τη δέουσα σοβαρότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο σκιώδης συγγετής, ο κύριος Λίσεκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή του κύριο Μποβέ. Στην ε, γνωμοδότηση αναφέρεται ο καρκίνος δικαίωσης σε βασική αιτία θανάτου ε, στο χώρο απασχόλησης. Εδώ πρέπει να δράσουμε λοιπόν, δεν χωράει εμφιβολία. Αλλά το να θέσουμε τέτοιες ε, αρχές δεν ξέρω κατά πόσον ε, είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Καταρχάς, τα όρια αυτά δεν μπορούν να ορίζονται κατά αποκόπη για όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη διάφορα συστήματα σε ό,τι αφορά τι ενεργειακέ στιγμέ και δεν μπορούν να συγκριθούν. Και έτσι το βασικό είναι να υπάρχει το ίδιο επίπεδο προστασία. Δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε λοιπόν. Οι οριακέ τιμέ δεν μπορεί να είναι πάντα μηδενικέ. Αυτή η αρχή θα πρέπει πάντα να τηρείται. Κατά δεύτερον, οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζονται και σε μια εκτενή μελέτη αντικτύπου. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της ε, τουρισμού των οριακών τιμών σε ό,τι αφορά το τρίχλο εθιλένιο. Κοιτώντα την πρόταση του εισηγητή, βλέπουμε πόσο απέχει από την μελέτη εντεκτύπου. και οι επιστήμονες ε, του σχετικής επιτροπής, ε, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι των συμβουλευτικών σωμάτων για την ασφάλεια συνεργασία, προτείνουν τα 54,7 4 μιλιγκράμμ ως όριο. Κάτω από το όριο αυτό λοιπόν οι επιστήμονες δεν θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνο στην υγεία και επίσης το θεωρεί και ο οικονομικός κλάδος αυτό εφικτό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνει 44,7 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα ο εισηγητής προτείνει 3,3 και νομίζω ότι απέχει πάρα πολύ από την μελέτη που Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς ε, της καλύτερης ε, νομοθεσίας. Κατά τρίτον, στην αιτιολόγηση της γνωμοδότησης αναφέρονται τα προστατευτικά. Αλλά οι ουσίε αυτέ που αναφέρονται, εξ όσων γνωρίζω και εξ όσων με ενημέρωσαν, δεν χρησιμοποιούνται στα φυτοπροστατευτικά. Και επίση, ε, η οδηγία του 2009 αποκλεί και δεν επιτρέπει την εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά τέτοιων καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων ουσιών για τις ε, φυτοπροστατευτικές ουσίες. Είναι πολύ περιορισμένη χρήση τους και οι Γερμανοί ειδικοί και εκπρόσωποι του κλάδου δεν πιστεύουν ότι υπάρχει έκθεση σε τέτοιες ουσίες. Ο καρκίνος του δέρματος αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αγροτών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι άλλωστε και το φως του ηλίου. Γιατί ο καρκίνος του δέρματος πολιτεί κυρίως αυτούς που εργάζονται έξω στον ήλιο, στον ύπεθρο και αυτό κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα ανά έτους και αυτό θα μπορούσε να αποτραπεί αν χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα μέτρα. Και εδώ στο σημείο θα ήθελα να πω και το εξή. Σήμερα στις 1 ε, στο Κοινοβούλιο, στο ASP, ε, ένα G στο μπαλκόνι, θα κάνουμε μια σχετική έκθεση και επί δύο ημέρες θα παρουσιάσουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους ένα δωρεάν έλεγχο ε, του δέρματος. Όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν μπορούν να περάσουν αν θέλουν για να κάνουμε και κάτι για την υγεία μας και για να επισημάνουμε το τι σημαντικό πρόβλημα είναι ο καρκίνος του δέρματος και πόσο μεγάλες μεταλλάξεις ενδεχομένω προκαλεί και θα καταθέσουμε τροπολογίες στην έκθεση του κυρίου Μποβέ και ελπίζω να μπορέσουμε με επικοδομητικό τρόπο να καταλήξουμε σε συμβασμούς ε, σωστούς και λογικούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Καδέμπαχ. Yeah, Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, 56 ε, έως 100.000 θάνατοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να κάνουν με εργαζόμενους και την έκθεση τους σε καρκινογόνες ουσίες κάθε χρόνο. 20... 20, 20 σε σχέση με τους υπόλοιπους θανάτους ε, στο χώρο εργασίας. Καλώ ορίζουμε λοιπόν αυτή τη νέα πρόταση για οριακές τιμές ε, σε ό,τι αφορά την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό αποτελεί άλλωστε εδώ και χρόνια έτοιμα πάγιο των ενώσεων εργαζομένων, προκειμένου να είναι δεσμευτικοί αυτοί οι όροι και να υπάρχουν και ελάχιστα όρια. Και χαίρομαι που η Επιτροπή Τάισεν ανακοίνωσε ότι το 2016 επρόκειτο να προτείνει οριακές τιμές για 16 έως και 50 τέτοιες ουσίες μέχρι το 2020. Διαπιστώνουμε ότι το 2016 εκδόθηκαν οριακές τιμές για 13 ουσίες και τώρα θα προσταθούν και περαιτέρω ουσίες για να καλύψουμε το κενό που μένει μέχρι τις 25 ουσίες που προβλέπονται στην οδηγία για τις καρκινογόνες ουσίες και να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία. Και τώρα δεν μιλάμε μόνο για γραφειοκρατικές αποφάσεις. Εδώ μιλάμε για θέματα ζωής ή θανάτου, ζωή ε, των ανθρώπων και για θέματα καλή ε, ποιότητας ζωής. Καλώ ορίζω λοιπόν την πρόταση και όπως αναφέρεται στην ετολογική σκέψη 15 πρέπει να μπουν και ανάλογε σκέψει και στην αντιδεκτικό του κειμένου. Και γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάντω τον συνάδελφο Μποβέ για την καλή του πρόταση για τις πιο πολλές μεμονωμένες ουσίες δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ μέχρι και αλλά να, να πω δύο λόγια για το τρίγλωριο εθλενείο. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να συμφωνήσω με τον εισηγητή για το ότι θα πρέπει να υπάρξουν διαφορετικές οριακές τιμές και χαίρομαι που ο σημείο αναφοράς ε, λαμβάνει την τιμή που ισχύει στην Αυστρία, τη χώρα μου. Και θα ισχύσει και στη Γερμανία συντόμως. θα γίνουν σχετικέ ε, μελέτε και έρευνε για την ε, μείωση τη οριακή τιμή αυτή και το, σε ό,τι αφορά την επαφή και την έκθεση σε καρκίνογόνε ουσίες ε, και την εκδήλωση τη ασθένεια μπορεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει 30 και 50 χρόνια και θα θυμάστε μια ουσία που χρησιμοποιούνταν πριν από πολλά χρόνια το τριχλωροετυλένιο, το οποίο και προκαλεί νόσους των νεφρών. Η εκτίμηση λοιπόν ότι η ουσία αυτή μπορεί να έχει όρια ασφαλή θεωρείται πλέον πεπηρεασμένη από 6 ppm θεωρείται ότι δεν είναι καρκινογενή η επίδραση στα νεφρά. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί σε χαμηλότερο επίπεδο λοιπόν από το προτινόμενο 10 ppm. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι συμφωνεί με την προδοσία αυτή, γιατί στην αντιλογική σκέψη 7 αναφέρεται ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη μείωση τη οριακή τιμή. και θα ήθελα να συμφωνήσω με ένα στοιχείο από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό το γεγονό ότι στο σημείο αυτό ο συνάδελφο Μπούφε αναφέρθηκε στην προστασία των γεωργών, γιατί πραγματικά θα πρέπει να προστατευθούν. Σε ό,τι αφορά την ηλιακή εκνοβολία, για παράδειγμα, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί πραγματική απειλή για την εργασία στην Ήπετρο και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αποτελεί αυτό υποχρέωση του εργοδότη και σε ό,τι αφορά την εργασία στα χωράφια να δίνει προστασία, να φροντίζει για την προστασία των εργαζομένων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν ε, στο σημείο αυτό να καταθέσουμε σχετικέ τροπολογίε. Μία ερώτηση θα ήθελα να απευθύνω γενικά για την κατάρτιση τη γνωμοτοτησή του συναδέλφου Μποβέ. <coughs> Γιατί εξαιρούνται οι υπάλληλοι οικιακοί υπάλληλοι. Ε, ρητά από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία ε, δεν υπάρχει κάποια σαφή ε, αιτιολόγηση για το γεγονό ε, ότι εξαιρούνται οι οικιακοί βοηθοί ή οι απασχολούμενοι στι κατοικίε από το πεδίο εφαρμογή τη νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αλλά θα παρακαλούσα όσοι λαμβάνουν το λόγο να μην μιλούν περισσότερο από ό,τι στην αρχική του παρουσίαση ο μα. μας. μισή λεπτό καθένα παρακαλώ, όχι παραπάνω. Ο κύριος Άγνιου. Πάλι έχουμε πρόβλημα με τη γαλλική διερμηνία. Δεν ακούγεται. Okay, Μήπως ε, δεν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο στην καμπίνα. Μισέλ τι γίνεται, Μισελ. Ακούς. Ευχαριστώ, κύριο Σάγνιο. Ευχαριστώ. Ο Τζοζέ Μπουβέ θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που εύχεται όταν μιλάει για μείωση της έκθεσης των αγροτών και των εργαζομένων στην γεωργία στα καρκινογόνα. Γιατί πιο, πιο σημαντικό από τα καρκινογόνα είναι ε, η καφεΐνη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ε, σταματάνε, πίνουν τον καφέ τους ας πούμε και αυτό είναι τεράστιο καρκινογόνο. Ε, μετά πάνε στο pub το βράδυ, το πίνουν αλκοόλ και αυτό είναι καρκινογόνα ουσία. εάν θέλετε απαγόρευση, θα πρέπει να τους αφαιρέσετε κάθε, απαγόρευση, κάθε απόλαυση τη ζωή τους. Ε, και το φως, ναι, όντως, μερικές φορές μπορεί να δημιουργήσει καρκίνο του δέρματος, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι γεωργός για να πας καρκίνο του δέρματος. Εάν κοιτάξεις από τις απειλές, τους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι, γεωργοί, ε, μην ξεχνάτε ότι ε, υπάρχουν ας πούμε και οι διευθυντές, τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία πέφτουν από ψηλούς ορόφους ας πούμε, ε, το να σίγουρα επιτεθεί ένα βοηδές, ε, να ε, να σε πλήξει ηλεκτρικό σοκ, ας πούμε, να ε, καείς και τα λοιπά, ε, τοξικές ουσίες. Ε, θα πρέπει κάπου να μπει μια, μια τελεία και να υπάρξει μια ισορροπία σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. όλοι θα ήθελα να περιοριστείτε σε 1,5-2 λεπτά. 1,5 λεπτά κυριο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ Eh, eh, Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Μποβέ, για την έκθεσή του. Ε, τη συμμερίζουμε απόλυτα. Οι γεωργοί και οι εργαζόμενοι στη γεωργία εκτίθενται καθημερινά σε μια σειρά από κινδύνους ε, λόγω χημικών ουσιών που μερικές φορές κλείνει το μικρόφωνο του μιλητή στον επαγγελματικό τους χώρο, λοιπόν, το γεωργικό, η διαδερμική έκθεση ε, είναι μια πρώτη πηγή έκθεσης ε, κινδύνου ε, και μπορεί να πάρει κανείς καρκίνο από, αυτές, αυτή την έκθεση. Οι οριακές τιμές είναι πολύ διαφορετικές στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, για τις πέντε αυτές ουσίες ε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα όρια, τα οποία ούτω ή άλλω είναι αρκετά ψηλά ε, σε ορισμένε χώρε, όπως στη Δανία, στη Γερμανία και στι κάτω χώρε. Ε, συγγνώμη, σε αυτέ τις τρει χώρες έχουν υιοθετηθεί καλύτερε πρακτικές. Ε, η οδηγία 37 του 2004 είναι ένα από τα βασικά κείμενα για την ε, προστασία της υγείας ε, στην εργασία. Όμως για τους ε, γεωργούς και τους εργαζόμενους στην γεωργία δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη από αυτή την οδηγία. Είναι σημαντικό λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας να, μπούμε και τους να μπουν και οι επαγγελματικοί χρήστες, που είναι ποιοι οι γεωργοί. γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε το κείμενο και θα υποβάλουμε και τροπολογίες και ευχαριστούμε τον κύριο Μποβέ. Ο κύριος Ντόρφμαν. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και σας ευχαριστώ και για τη σημερινή συζήτηση. Ο καρκίνος είναι σημαντικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί πολλοί ετικήσονται στην ασθένεια αυτή και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και ποιε είναι οι συνδυαστικοί παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως να επιδρούν και οι οποίοι δεν είναι ξεκάθαροι. Τι θα πρέπει λοιπόν να γίνει για να τα αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα πρέπει να τα πάρουμε στο σοβαρά το θέμα. Κάποιε χώρε σημειώνουν πρόοδο και αυτό είναι πολύ θετικό. Και ω εκπρόσωπο τη Δανία, εγώ ξέρω ότι είναι κάτι στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα η ασφάλεια στον χώρο εργασία. Αλλά όπω είπαν και άλλοι, όταν κανεί ε, δουλεύει έξω, εκτίθεται σε σκόνη και ήλιο, ενδεχομένω να διατρέχει κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μακροπρόθεσμα. Και ξέρουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ε, όταν ε, κατασκευάζονται στάβλοι, για παράδειγμα, ή ε, τα υλικά για την στέγη μπορεί να περιλαμβάνουν καρκινογόνες ουσίες. Και επίσης έχω υπόψη μου και τα εργαλεία. Όταν κανείς ψεκάζει. Πώς ξέρει, για παράδειγμα, αν τα εργαλεία είναι παλιά, πέντε χρονών, για παράδειγμα, και ε, διατραχεί κίνδυνο μέσω αυτών. Έτσι λοιπόν στην ε, Δανία έχουμε εισαγάγει υποχρέωση ελέγχου, περιοδικού ελέγχου των ε, μηχανημάτων και των εργαλείων, όπως για παράδειγμα τα οχήματα. Έτσι λοιπόν σκοπεύουμε να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Δενανό. Ευχαριστώ. Όντως ενδιαφέρουσα συζήτηση και έχουμε καθήκον εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προστατεύσουμε τους καταναλωτές μεν, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και αυτούς που εφοδιάζουν τους καταναλωτές με τρόφιμα, τους γεωργούς δηλαδή. Είχαμε πολύ άριθμα παραδείγματα στο παρελθόν ε, στους ε, καλλιεργητές οποροφόρων ε, παραγωγούς λαχανικών για ολέθρια αποτελέσματα για τους ίδιους Γιώργους, τις οικογένειές τους και το περιβάλλον. Οπότε δεν λέω ότι θα πρέπει με τα ξερά να κάψουμε και τα χλωρά, αλλά να είμαστε προσεκτικοί και να λάβουμε τα μέτρα μας. Και είναι πολύ εύστοχη και αξιόλογη η γνωμοδότηση του κυρίου Μποβέ. Χρειαζόμαστε και κάποια ευρωπαϊκά μέτρα για τις οριακές τιμές για κάποιες χημικές ουσίες. Οπότε το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε την παραγωγή, αλλά να συνεχίσουμε την παραγωγή υπό ικανοποιητικές συνθήκες και για τους γεωργούς και για τους καταναλωτές. Έχουμε προϊόντα όπως το τρίχλωροεθυλένιο ή όλα τα προϊόντα από βενζίνη ή βενζένιο. Οι πτυτικές ενώσεις του βενζονίου που έχουν αποκριθεί επικίνδυνα. Δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλους αυτούς τους κινδύνους ε, οι γεωργοί, γιατί οι καρκινογόνες ουσίες ε, φέρουν αποτελέσματα μακροπρόθεσμα, οπότε θα πρέπει να έχουμε και μακροπρόθεσμη προοπτική. Και ευχαριστώ τον Ζωζέ Μποβέ για την έκθεση του κυρία Μίλλερ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα εξ ονόματο ε, τη ε, σκιώδους εισηγητριάς μας να πάρω το λόγο. Διαβάσαμε λοιπόν την πρόταση του κυρίου Μποβέ και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ θετικό το γεγονό ότι συμπεριλαμβάνονται στο σημείο αυτό και η Γεωργία Και μιλάμε για 22 εκατομμύρια ανθρώπους άλλωστε, οι οποίοι πραγματικά μπορούν να προστατευτούν τον τρόπο αυτό από την έκθεση σε καρκινογόνες ουσίες και για τις οριακές τιμές. τιμές. Ασφαλώς θα πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή. Ξέρω ότι η Γερμανία από το 2018 θα ρίξει τις τιμές στα 3,3 μιλιγκράμμ σε ό,τι αφορά το χλωρό εθιλένιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη οι διαφορές όμως που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την έκθεση στην ουσία αυτή. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το ότι μειώνεται η οριακή τιμή στο σημείο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δοθεί ένα έναυσμα σε ό,τι αφορά την προστασία της υγείας. Και ο έλεγχος των οριακών τιμών από μόνος του αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα σε ό,τι αφορά και ενδεχόμενη μείωση της οριακής αυτής τιμής. Το κατά πόσο στο σημείο αυτό θα συμπεριληφθούν ρητά και τα φυτά προστατευτικά στοιχεία, οι ουσίες αυτές οι οποίες ε, όντως ρητά εξαιρούνται, δεν ε, είμαι σίγουρη ότι χρειάζονται. Θα συμφωνήσω με τον ε, συνάδελφο Γκίζε και θα το εξετάσουμε και και παρόλα αυτά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την γνωμοδοτησία. Αυτά τα τρία κριτήρια αυτά μα βρίσκουν σύμφωνο. Ευχαριστώ κύριο Μπούντα. Σας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνικός. Είναι χρήσιμες τέτοιες συζητήσεις για την προστασία των εργαζομένων και την επέκταση της προστασίας όλων των απασχολουμένων στον κλάδο από καρκινογόνες ουσίες. Τι είναι όμως καρκινογόνος ουσία? γιατί οποιαδήποτε ουσία που χρησιμοποιείται υπερβολικά μπορεί να προκαλέσει ασθένειες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ανάγκη έχουν τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου και διάγνωσης ε, των καρκίνων στον γεωργικό πληθυσμό γιατί πολλοί αγρότες σε απομονωμένες περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτική ιατροφαρμακευτική και υπηρεσία υγείας. Θέλουμε λοιπόν μηχανισμούς διάγνωσης του καρκίνου και στην Ήπεθρο για να γίνεται έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος και άλλων μορφών καρκίνου. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω στον εισηγητή ότι προφανώς συμφωνώ ότι οι εργαζόμενοι στη γεωργία, οι γεωργοί, όλοι όσοι ασχολούνται τόσο πάντων με φυτοϊγειονομικά προϊόντα, προφανώς θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερο έλεγχο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια οδηγία βέβαια, όπου αφορά τους γεωργούς καθώς και τους επαγγελματίες στη γεωργία. Ε, ο κάθε ένας από αυτούς που χειρίζονται τα φυτογενομικά προϊόντα θα πρέπει να έχει ε, ένα πιστοποιητικό για να μπορεί να τα χειρίζεται. Μιλάω και για τους γεωργούς και για τους ε, επαγγελματίες στον χώρο της γεωργίας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν μια κατάρτιση για τη χρήση αυτών των προϊόντων. θα πρέπει να κάνουμε ίσως ε, κάποιες τροποποίησεις, ούτω ώστε να έχουν καλύτερη κατάρτιση και οι γεωργοί και οι επαγγελματίες στον χώρο της ε, γεωργίας, τέλο πάντων όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα προϊόντα, κατάρτιση για τη χρήση τους. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε αυτό το στοιχείο της ε, κατάρτισης να το εντάξουμε και το θέμα της πιστοποίησης επίσης των ανθρώπων αυτών να το εντάξουμε στα κείμενα. Ο κύριος Φλάνακαν, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα συμφωνήσω με πολλά από αυτά που δήλωσε ο εισηγητής και καλωσορίζω την όλη ιδέα της επέκτασης για να καλυφθούν πιο πολλοί εργαζόμενοι. Θα έχω και εγώ μια παρόμοια ερώτηση με αυτή που τέθηκε προηγουμένω. Γιατί δεν περιλαμβάνονται εκεί, εκεί οι υπάλληλοι. Και επίση, σχέση με αυτά που είπε ο κύριο Αγνιό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα αυτά που ανέφερε είναι καρκινογόνα, αλλά ε, φέρνουν και απόλαυση και οι ενδορφίνες που προκύπτουν μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου. Δεν βλέπω ότι απόλαυση υπάρχει από το να εκτίθεται κανείς σε καρκινογούνες ουσίες ε, και σε υψηλές ε, οριακές τιμές. Δεν υπάρχει καμία απόλαυση, δεν υπάρχει καμία επιβράβευση αν θέλετε. Και νομίζω ότι όπως συχνά σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες για την υγεία, σημαντικό είναι να μειώσουμε τις ανησυχίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την επεξεργασία τεχνικών ζητημάτων και χημικών ουσιών. Άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με την γλυφοσάτη και το οποίο είναι ακόμα εκρεμές του τι είναι επικίνδυνο και τι δεν είναι επικίνδυνο και αυτό με οδηγεί στην ε, επεξήγηση της τη από την έψη που είχε έρθει εδώ. Ένα πράγμα είναι σαφέ ότι είμαστε περιορισμένοι και πάντα θα είμαστε περιορισμένοι όσο δεν έχουμε ανεξάρτητη α, παροχή συμβουλών για τα χημικά αυτά. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, γιατί πού να βρει κανεί τα δισεκατομμύρια να τα εξετάσει όλα αυτά τα στοιχεία, όλε αυτέ τι ουσίε. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονό. όσο δύσκολο και αν είναι να αποφασίσουμε ανεξάρτητα το τι είναι ασφαλές και τι δεν είναι ασφαλές. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Τώρα το πώς θα το πετύχουμε είναι μια διαφορετική ιστορία βέβαια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλιν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ζωζέ Μποβέ και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κ. Ζαγκίζη και γιατί δεν καταλαβαίνω απόλυτα αυτά που είπε, ότι εμείς δηλαδή ω πολιτικοί δεν θα έπρεπε να ξεκινήσουμε συζήτηση για τις συριακές τιμέ, Μα αν δεν ξεκινήσουμε εμείς τη συζήτηση αυτή, ποιο θα το κάνει, Ποιο άλλο θα το κάνει. Αναφέρθηκε ότι στη Γερμανία είναι διαφορετικέ οι οριακέ τιμέ, ε, αλλά στο ό,τι αφορά το τρίχλωρο εθιλένιο, η Γερμανία είναι αυτή που έθεσε την οριακή τιμή το 2018. Γιατί δεν καταλαβαίνω, λέτε, ότι δεν θα πρέπει η Ευρώπη να προσαρμοστεί στι οριακέ αυτέ τιμέ. Είναι λογικό το ότι υπάρχουν διαφορετικέ οριακέ τιμέ και θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι βέλτιστε πρακτικέ. Και οι αγρότες ε, Ρωτήσατε δηλαδή την, Ευρω... την Γερμανική Ένωση Ακροτών και σας είπαν ότι δεν υπάρχουν ε, φυτοπροστατευτικά που προκαλούν ε, καρκίνο. Τι σημασία έχει αυτό. Για την πρόληψη και την προστασία της ε, υγείας των αγροτών θα έπρεπε να κάνουμε κάποια προσπάθεια δεν αρκεί αυτή η δήλωση ότι κατά τη γνώμη του δηλαδή δεν υπάρχουν καρκινογόνε τέτοιε ουσίε. Θα ήθελα λοιπόν να σα καλέσω να αναθεωρήσετε την απόψη σα. Γιατί νομίζω ότι κινείται πάρα πολύ προ την κατεύθυνση της, ε, των αγροτικών ενώσεων και τη ε, χημική βιομηχανία η άποψή σα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Πόλτσακ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τα περισσότερα τα καλύψαμε. Θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω το υπόβαθρο της πρότασης, γιατί προστίθεται μια νέα νομική βάση με κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για το άρθρο 153 της συνθήκης, που ισχύει μόνο στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς. Οπότε από νομική άποψη δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε άλλο παρά μόνο στους εργαζόμενους, στους μισθωτούς, όπως προσδιορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη, στα θέματα των κοινωνικών υποθέσεων ε, προσδιορίζουμε κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, ελάχιστους όρους. Είναι σαφές το μήνυμα, υπάρχει επικουρικότητα στην περίπτωση αυτή. Δεν ε, έχουμε ε, διατάξεις όπως τις ενίας αγοράς όπου έχουμε μία οριακή τιμή και ένα κανονισμό. Εδώ προβλέπουμε ελάχιστες οριακές τιμές. Και λέμε, όταν ένα κράτος μέλος ε, δύναται, όταν επιθυμεί μπορεί να βελτιώσει τις τιμές. Αλλά εμείς θέτουμε το κατώτατο όριο. Και με βάση τη νομική αυτή βάση υπάρχει υποχρέωση διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου που μπορούν να διαπραγματευτούν και ειδικέ συμφωνίες που μετά να, μεταφερθούν στην νομοθεσία. Αυτή είναι η τυπική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα καρκινογόνα, τι καρκινογόνες ουσίες που εγκρίθηκε με βάση αυτή τη νομική βάση, προβλέπει διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου, αλλά διαβούλευση και με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασία. Είναι τριμερή αυτή η Επιτροπή σε όλα τα κράτη-μέλη έχουμε τους ε, βασικούς εργοδότες και τα βασικά συνδικάτα που συμμετέχουν σε αυτή την τριμερή συμβουλευτική επιτροπή. Γιατί όταν ασχολούμαστε με θέματα ασφάλειας και υγείας θέλουμε να εμπλέκουμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να εξασφαλίσουμε και εφαρμογή των ηλυμένων μέτρων. Και ο τρόπος που υποβάλαμε την πρόταση είναι ε, καταρχήν ζητήσαμε επιστημονικές ε, συμβουλές και πορίσματα από πολλές πηγές τις υποβάλαμε στην Επιτροπή και αυτά τα τρία μέρη εξέτασαν τις οριακές τιμές από την επιστημονική σκοπιά και κα, κατέληξαν στις συγκεκριμένες προτάσεις για τις οριακές τιμές. Κατόπιν η Επιτροπή έλαβε την πολιτική απόφαση να μην τροποποιήσει τις οριακές τιμές που προέκυψαν αυτή την τριμερή συζήτηση μεταξύ εργοδοτών, κρατών μελών και συνδικάτων. Μάλιστα συντάξαμε και μελέτη επιπτώσεων για να διαπιστώσουμε ε, αν υπάρχουν ε, ανεπιθύμητα αποτελέσματα κάτι που ξέφυγε από τους εταίρους δηλαδή, ε, δηλαδή και επιβεβαιώθηκε η έλλειψη τέτοιων αρνητικών ανεπιθύμητων συνεπειών. Όπως είπα, η πρόταση αποτελεί τμήμα μια σειράς προτάσεων που ε, έπρεπε να είχαν υποβληθεί πέρυσι, θα υποβληθούν και φέτος και θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια. Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση αυτή την προηγούμενη εβδομάδα και ενέκρινε όλες τις οριακές τιμές αμετάβλητες με ελάχιστες τεχνικές τροποποίησεις. Το επιχείρημα του Συμβουλίου είναι να μην αποκλίνουμε από τη συμφωνία στην Τριμερή Επιτροπή. βέβαια, αν η απόκληση είναι σημαντική, θα επηρεάσει και τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Γι' αυτό και εσείς να μην αποκλίνουμε ιδιαίτερως από την συμφωνία αυτή των ενδιαφερομένων. Αυτά δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Αν δεν κάνω λάθος, ανέκυψε και ένα άλλο θέμα, παρόλο που δεν είμαι ειδικό για τα θέματα, εγώ ασχολούμαι με το ζήτημα της απασχόλησης. Αναφερθήκατε στα φυτοφάρμακα, στα εντομοκτώνα. Οι, τα καρκινογόνες ουσίες του 1α δεν εγκρίνονται ως φυτοφάρμακα. Αυτόματα αποκλείονται από τα φυτοφάρμακα, από τις φυτοπροστατευτικές ουσίες. Αυτό ήταν το τεχνικό ζήτημα. Αλλά δεν είμαι ειδικό για τα θέματα αυτά και δεν μπορώ να αναπτύξω πιο διεξοδικά αυτό το σημείο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η συγγετής μας τώρα, ο κύριος Μποβέ. Δεν θα επανέλθω σε όλα τα θέματα, θέλω να σχολιάσω όμως ένα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν το κατάλαβαν και το συζήτησαν πάρα πολύ. Δεν το κατάλαβαν, ας πούμε. Υπήρχε στο κείμενο στην τροπολογία 3, εκεί που μιλάω για τους εργαζόμενους με την εξαίρεση των ε, οικιακών βοηθών ε, που απασχολεί ένα ε, εργοδότης, αυτός ο ορισμός δεν είναι δικός μου. Προέρχεται από το κείμενο ε, της οδηγίας υγεία και ασφάλεια 89 391. Από εκεί την πήρα και εκεί προσθέτω και, την, ε, και τον ορισμό της οδηγίας 11.07 του 2009 ε, για τους γεωργούς. Ε, και έτσι μπορούμε να, να καλύψουμε το σύνολο των χρηστών με αυτές τις δύο οδηγίες. Δεν έβαλα εγώ αυτή την έννοια των οικιακών βοηθών, δεν ξέρω από πού προέρχονται. Στο παρελθόν, όταν είχαμε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, μιλήσαμε για αυτούς. Φυσικά δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε διακρίσεις τέτοιου τύπου, όπως είπαν κάποιοι, απλώς χρησιμοποίησα τους όρους των κειμένων που έχουμε, των δύο οδηγιών. Ίσως ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Κοινωνική Επιτροπή για να τροποποιήσουμε αυτό το κύμα που μοιάζει λίγο απαρχιωμένο. Αυτό ήθελα να σας απαντήσω, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ακούγοντας όμως την Κομισιόν, βλέπω ότι υπάρχει διαφωνία και το θέμα της υγείας για μένα είναι ουσιαστικό θέμα και το θέμα των κατοφλίων είναι ουσιώδες ούτω ώστε να υπάρξει πρόοδος ε, στην καταπολέμηση του καρκίνου και της έκθεση των προσώπων στο χώρο εργασίας. Βάζοντας, παίρνοντας την μέγιστη επιτρεπόμενη δόση ε, στη χώρα που έχει τους πιο αυστηρούς κανόνες ε, και κρατώντας το όσα αναφορά, νομίζω ένα, ένα μήνυμα θετικό που δίνουμε σε όλες τις χώρες. Ε, η Αυστρία ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά για το τρίχλωρο και η Γερμανία αποφάσισε να την ακολουθήσει. Είναι λοιπόν αυτό ένα πολύ καλό βήμα. Προς εκεί πρέπει να κινηθούμε και να βοηθήσουμε τις χώρε ούτω ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και τους ε, γεωργούς με τον ίδιο τρόπο. Και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Ε, αυτό το, αυτή την απόχρωση, αυτό το νόημα ήθελα να δώσω στο κείμενό μου. Σας ευχαριστούμε. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει 26 Ιουνίου, μία το μεσημέρι. Η έγκριση της έκθεσης θα γίνει τον Οκτώβριο ε, και στην αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόλησης, τον Νοέμβριο. Ε, και ε, καθορίζεται εδώ και είναι συγκεκριμένος μάλλον και ο ρόλος των παραγωγών αυτών των ουσιών. Περάμε στο επόμενο θέμα. την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης. Συντάκτης γνωμοδότης είναι ο κύριος Γιένς Ρόντε. Αρμόδια καθήλια επιτροπή με βάση το άρθρο 55 είναι δύο επιτροπές, οι επιτροπές περιβάλλοντος και η επιτροπή ε, και βιομηχανίας. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ρόντε, για να μας κάνει την εισαγωγή. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να φύγω. Ψηφίζουμε στη νομική επιτροπή. Η και θα καταγράψει προσεκτικά τα σχόλιά σας και θα μου τα διαβιβάσει για να τα λάβω υπόψη. Λυπούμε, αλλά πρέπει να φύγω σε λίγο. Θα ήθελα πρώτα να χαιρετήσω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει μια συντονισμένη και συνεκτική εφαρμογή των νομικών, οικονομικών και στρατηγικών σκοπών και στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ανάπτυξη μιας διακυβέρνησης Ενεργειακής Ένωσης είναι να εξασφαλίσουμε ε, υλοποίηση των στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ενωσιακό επίπεδο και να γίνει και παράδειγμα προς και για άλλους κλάδους. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία ειδικά, η πρόταση προβλέπει υποχρεώσεις ε, ενημέρωσης των κρατών μελών, υποβολής εκθέσεων για τη δική του στρατηγική για μείωση των εκπομπών, για, τις, ε, για τα μέτρα τους και τα θέματα αποσύρσεων σε, στον, Ευρω... στον γεωργικό τομέα και επίσης το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιοκαυσίμων που ε, παράγονται από τις βασικές αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, ε, ε, πρόθεση μέτρων ώστε να προωθηθούν μέτρα για τη βιομάζα, ακόμη και τη βιομάζα του γεωργικού τομέα και ενεργειακή κατανάλωση από μεμονωμένους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της γεωργίας. Πρότεινα κάποιε ατροπολογίε κυρίω τεχνική υφή, μερικέ φορέ αφορούν προσαρμογή τη διατύπωση. Για παράδειγμα, στα πλαίσια τη ε, υποβολή εκθέσεων για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει σαφεί κατευθυντήριε γραμμέ για τα κράτη-μέλη για την υποβολή εκθέσεων για τη βιοενέργεια. Επίση, ε, ε, αν καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ένα κράτο μέλο δεν έχει συντελέσει επαρκή πρόοδο ό,τι αφορά του στόχου υλοποίηση των μέτρων, όπω προβλέπει το, το εθνικό σχέδιο το ενεργειακό και το του κλίματος θα μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένες απαιτήσει και προϋποθέσεις για το κράτος μέλος. Και αυτές οι προϋποθέσεις αντικαθιστούν το σύστημα των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το ενδιαφερόμενο κράτος. Γιατί οι συστάσεις, επειδή δεν είναι δεσμευτικές, δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές στην περίπτωση αυτή και μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω επανεθνικοποίηση. Κάτι που δεν μας βρίσκει σύμφωνο. Θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση τη γεωργικής μας πολιτική. Στι 27 ε, Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τις τροπολογίε και 30 Αυγούστου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η υιοθέτηση ενός κειμένου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ε, είναι επίγουσα, ούτω ώστε να προωθηθούν οι πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια ε, με ορίζοντα το 2030. Η Γεωργία παίζει στρατηγικό ρόλο και για τη μείωση των εκπομπών καθώς και για την αύξηση της απορρόφησης με σκοπό το, την υλοποίηση των εθνικών στόχων ε, και την πρόθεση των, α, της για τις ανανεώσιμες ενέργειες καθώς και των ενεργειών που παράγονται από τη βιομάζα. Η θέση των, ε, του εισηγητή τη συμμεριζόμαστε, όμως η Μικέλα Τζουφρίντα που είναι η σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μας την οποία την καθιστώ, λέει ότι πρέπει να επιμείνουμε σε κάποια στοιχεία. Καταρχάς, το πρώτο, για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στις, ε, στην επικοινωνία μεταξύ κομισιών και κρατών μελών, οι συστάσει ή οι συγκεκριμένε προποθέσει ανά χώρα θα πρέπει να είναι δημόσιε. Επίση, θα πρέπει να είναι γνωστά και δημόσια τα κριτήρια καθώ και οι δείχτες που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για την αξιοποίηση των εθνικών και ε, αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων. Εν συνεχεία, πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερο προβληματισμό και σκέψη για το άρθρο 13. Το άρθρο 13 με το οποίο η Κομισιόν λέει ότι ένα κράτο μπορεί να ξαναδεί να επικαιροποιήσει το εθνικό του σχέδιο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο μόνο για να καθορίσει πιο φιλόδοξου ε, στόχου και όχι αλλιώ συμφωνούμε με αυτή τη διάταξη, αλλά όμω έχουμε και κάποιε αμφιβολίε. Γιατί καταρχά αυτό ο κανόνα δεν αφήνει περιθώριο στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τι πολιτικέ του με βάση ε, το πλαίσιο στο οποίο ισχύει και την πραγματικότητά του. Ή ε, επίση δημιουργεί ένα στρεβλωτικό μηχανισμό. Δηλαδή το κράτο μέλο το οποίο δεν ξέρει να γυρίσει προ τα πίσω μπορεί να, να θέσει ε, στόχου πάρα πολύ χαμηλού και καθόλου φιλόδοξου. Επίση, η διακυβέρνηση ε, προβλέπει στο 27 μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα χρηματοδότηση που ε, προωθεί ε, έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Καλή είναι, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Επίσης, τεράστια σημασία έχει η γεωργία, για τη γεωργία έχουν τα παρατήματα. Τα παρατήματα όπου ορίζονται τα θέματα που συνδέονται με τη γεωργία και που εντάσσονται στα εθνικά σχέδια και καθορίζονται σε σχέση, ε, στα πλαίσια της επικοινωνίας κρατών μελών με την ε, Κομισιόν. Αυτό συνδέεται με άλλα, ε, με άλλα ντοσιέ τα οποία είναι ανοιχτά, όπως παραδείγματος χάρη το LULUCF η χρήση γη, αλλαγή γη κτλ. ή ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Οι τροπολογίε ακριβώ λοιπόν θα πάνε προ αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή να υπάρξει μια εναρμόνιση με αυτά που καθορίζουν οι άλλοι κανονισμοί, LULUCF κτλ. Χωρί βεβαίω να στραβλώσουμε την πρόταση τη Κομισιόν. Αλλά να τονίσουμε ότι η Γεωργία πρέπει να έχει ειδικό ρόλο στην ε, διακυβέρνηση και στη διαμόρφωση, συγγνώμη, στην διαμόρφωση της ε, διακυβέρνησης. Ευχαριστώ κύριο Σκάρθη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ εν πολύ με τον κύριο Δεκάστρο. Και ο συνδυασμό ε, των κανονισμών και των οδηγιών είναι καλή πρακτική και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε απλούστευση. Αλλά δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μαζική εκχώρηση εξουσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει αυτός ο συνδυασμός ε, να έχει άλλο στόχο. Μετά τις, δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση της Ενεργειακής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε ε, διαπιστώσει. Μία πολιτική που ε, ευνοεί τις πολυεθνικές εταιρείε εις βάρος ε, των επιμέρους κλάδων, οι οποίοι υποφέρουν από τη γραφειοκρατία. Και μάλιστα ε, δεν τηρούνται ούτε οι αρχές επικουρικότητας και αναλογικότητας ούτε επαρκή ε, συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση των εθνικών σχεδίων, ούτε γίνονται επαρκεί διαβουλεύσει σε εθνικό επίπεδο. Και μάλιστα αυτό το σήμα κινδύνου έστειλαν έξι κοινοβούλια προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει λοιπόν γενική αποδοχή των προτάσεων ε, γιατί μερικές φορές επεμβαίνει σε εθνικές πολιτικές ε, για την ενεργειακή πολιτική δεν θα πρέπει με μια νέα ενεργειακή πολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύει τις πολυεθνικές ε, που η θέση τους είναι ήδη προβληματική. Πάντως ε, προσβλέπω σε συνέχιση το συζητήσω με τους υπόλοιπους ε, σκιώδης ηγητές και θα καταθέσουμε τροπολογία στην Επιτροπή για να αμβλύνουμε τις πιο αρνητικές πτυχές και να προβάλλουμε τις ανάγκες των γεωργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέροντας στο επίκεντρο των συζητήσεων. Κυρία Σκότ, Χαίρομαι που έχει γνωμοδότηση άγρη για τι προτάσει για την Ενεργειακή Ένωση, γιατί είναι σημαντικό να συνδέσουμε τη γεωργία, το κλίμα και την ενέργεια. Ε, και εμεί ε, μπορέσαμε να το κάνουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Η Συμφωνία του Παρισιού θέτει στόχου για τη μείωση των εκπομπών του διοξείδου άνθρακα, αλλά κυρίω αφορούν την ε, βιομηχανία. Και έχουμε καλά νέα ότι απορρέουν επενδύσει, άρα έχουμε κάποια σημεία πρόοδου. Αλλά δεν αρκούν αυτά για το κλειό. Αυτά που κάνουμε για τη βιομηχανία, δεν μπορούμε, με αυτά δεν μπορούμε, να, να πετύχουμε το στόχο του να σταθούμε στο 2,5%, να μειώσουμε δηλαδή το, τη θερμοκρασία, να μην αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από το 2,5 βαθμούς. Πρέπει να κάνουμε κάποιες ε, προσπάθειες για τα βιοκαύσιμα κτλ. Αλλά αφορούν κυρίως ε, το φινικέλαιο και την εισαγωγή του ε, φινικελίου και μερικές φορές μάλιστα αυξάνουν και τις εκπομπές αυτά τα βιοκαύσιμα. Επομένως, ε, πρέπει να κρατήσουμε τη σχέση μας με την, ε, ανάμεσα στο κλίμα και στο έδαφος, που είναι σημαντικό. Και οι πέντε στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης είναι πολύ σημαντικοί για τη γεωργία. Καταρχάς, η ενεργειακή ε, ασφάλεια, η αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε ε, Εθνικέ προσπάθειες μέσω της υδρογρομάτιση κτλ. Ε, αν προτείνουμε τα βιοκαύσιμα θα πρέπει αυτά να πληρούν τι ανα, αναγκαίες προϋποθέσεις. Να μειώσουν δηλαδή πραγματικά το διοξείδιο του άνθρακα ε, και επίσης να μην ε, ξεχνάμε και τα τρόφιμα που πετιούνται κτλ. Επίσης να έχουμε μέτρα για να επιτρέψουμε καύσιμα μόνο αν, από το εξωτερικό μόνο ή μάλλον να μην επιτρέψουμε ε, να εισάγονται καύσιμα σε χαμηλέ τιμέ αν έχουν ε, πολύ μεγάλη περιβαλλοντική επίπτωση. Επίσης ε, θα πρέπει ε, όλους τους, ε, τους τομείς μεμονωμένα να τους δούμε ε, στην κατανάλωση ενέργειάς τους. για την μείωση των εκπομπών και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ε, θα το δω αυτό προσεκτικά, για την έρευνα καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα υπάρχει τεράστιο δυναμικό καινοτομία. Αλλά θα πρέπει ε, να αντισταθμίσουμε, να δούμε από τη μία τις τεχνολογικές αλλαγές και από την άλλη την ανάγκη ε, για καινοτομία. Συμφωνώ με τις βάσεις της πρότασης του ε, εισηγητή, χρήσιμη αφετηρία. Ε, λέει ότι η Κομισιόν στα πλαίσια των εκθέσεων θα πρέπει να έχει να έχουν ε, κατευθυντήριες γραμμές σαφείς ε, και θα πρέπει να δούμε ε, και τις επιπτώσεις του διοξείδου του άνθρακα και τη μετατόπιση των εκπομπών. Θα πρέπει επίσης, αν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες παρεκκλήσεις, να, κάνουμε, να παίρνουμε μέτρα από την αρχή. γίνεται μια πρόταση ότι υπάρχουν, έχουν δυσκολίες τα, στα κράτη-μέλη να υποβάλουν εκθέσει για τη χρήση γη αλλαγή χρήση γη κτλ. ή τι τιμέ των προϊόντων. Ε, είναι δύσκολο να τα μετρήσουμε, βέβαια, αλλά να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και θα το συζητήσουμε αυτό στου ε, σκιώδει. Θέλω να το συζητήσουμε με τους άλλους σκιώδει. Περιμένω αυτή τη ε, συζήτηση και ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ο κύριος Γιάρ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το σχέδιο γνωμοδότησής του και για το ότι έφερε στο επίκεντρο της συζήτησης τη σχέση γεωργίας και κλιματικών αλλαγών. Για τη βιομάζα έχει γίνει σφοδρή συζήτηση. Γνωρίζουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των βιοκαυσίμων και ότι μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα. Τι συνέβη όμως εδώ. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι οι προθέσει μα ήταν αγαθές, αλλά τα αποτελέσματα δεν μας δικαίωσαν. Τι συνέβη λοιπόν. Με την ενεργειακή παραγωγή, που συνήθως γίνεται στη γεωργία, ε, ενώ είχε ξεκινήσει η ενεργειακή παραγωγή από τη γεωργία, πέρασε στην βιομηχανία μέσω της παραγωγής φινικελαίου ή χρησιμοποίησης άλλων πρώτων υλών θα πρέπει να έχουμε επιστοποιημένη βιομάζα με πολλαπλή συμμόρφωση, με οικολογικοποίηση και κάποιους βασικούς κανόνες για τους γεωργούς, γιατί δεν δίνουμε τη δέωσα προσοχή στη βιομάζα. Γιατί θα ξεφύγει από τον έλεγχό μας η βιομάζα αν επικεντρωθούμε μόνο σε εισαγόμενη βιομάζα. Σε πολλές αγροτικές περιοχές η παραγωγή της βιομάζας είναι η μοναδική ευκαιρία ε, μιας ε, ενεργειακής αυτάρκειας με φωτοβολταϊκά, με αιωλική ενέργεια, με τη χρήση των δασών, με καταστάσεις ε, βιοαερίου ή υπάρχουν περιοχές που ενώ ε, περιτριγυρίζονται από δάσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο και φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους. Είναι απαράδεκτο αυτό. Επίσης έχουμε τοπικές αρχές και μεγάλες ε, ε, επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη τοπικών δικτύων ε, παραγωγής ενέργειας. Είναι κρίμα γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία που την αφήνουμε να ανεκμετάλλευτη. Έτσι θα μπορούσαμε να παράγουμε βιώσιμη ενέργεια υπό τρόπο, να παράγουμε βιομάζα και να καταπολεμήσουμε ταυτόχρονα και τις κλιματικές αλλαγές. Παρακαλώ μην ξεχνάτε ε, κύριε Σιγητά και αυτή την πτυχή. Γιατί η Γεωργία μας δίνει μια ευκαιρία και όχι κίνδυνο για να παράγουμε ενέργεια με τέτοιο τρόπο. Ο κύριος Άγνιου. Ευχαριστώ. Η βασική εργασία των γεωργών είναι να παράγουν τρόφιμα. Μπορούν ως υποπροϊόν να παράγουν και ενέργεια, για παράδειγμα τα ζαχαρότευλα που πηγαίνουν σε εργοστάσια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, από το πολτό που δεν χρησιμοποιείται βιοεθανόλη. Βέβαια, θα μπορούσε αυτός ο πολτός από τα σαχαρότευτα να, να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή. Οπότε έχουμε μια πόλη. Το ίδιο ισχύει και για τα δημητριακά που κυρίω χρησιμοποιούνται ω τρόφιμο, αλλά το άχυρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω ενέργεια. Αν όμω το άχυρο το πάμε ε, από τη φάρμα στην βιομηχανική παραγωγή, ε, θα πρέπει να εισάγουμε για την ενέργεια για την φάρμα, οπότε και εκεί έχουμε απώλεια. Σίγουρα ε, έχουμε και σπατάλη στα τρόφιμα και κρίμα είναι να μην τα χρησιμοποιούμε και αυτά όταν, αντί να τα σπαταλούμε. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα όταν ε, η μοναδική εργασία του Γιώργου είναι αντί να παράγει τρόφιμα να παράγει ενέργεια. Αυτό γίνεται με, με την καλλιέργεια ραποσίτου για παράδειγμα και μάλιστα χρησιμοποιείται ο αραβόστος ως ενεργειακό προϊόν. Μετά πρέπει να γίνει όργωμα στο χωράφι και να καλλιεργηθεί και πάλι με αραβόστο για να παραχθεί και πάλι ενέργειο. Έχουμε λοιπόν και τα τρακτέρ που απορροφούν πολύ δίζελ χρειάζεται μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν, να μεταφερθούν σε μεγάλη απόσταση μέχρι το εργοστάσιο και εδώ έχουμε επίσης παραγωγή, ε, χρησιμοποίηση μάλλον, κατανάλωση μεγάλη καυσίμων. Ε, αυτό είναι πραγματικά σκάνδαλο τέτοιες πατάλες καυσίμων. Και μάλιστα εξαπλάσια ενέργεια χρειάζεται για την παραγωγή τέτοιων καλλιεργιών από ό,τι προσφέρουν ενέργεια. Οπότε σίγουρα χρειάζεται κάποια ενέργεια ο Γιώργος για να παράγει οικολογικές καλλιέργειες, αλλά και εδώ το οικολογικό λόμπι τον εμποδίζει, γιατί αν μπορούσε να χρησιμοποιεί γλυφοσάτη και γενετικό τροποποιημένους οργανισμούς θα μείωνε την κατανάλωση ενέργειας στην ε, φάρμα του. Όμως οι περιβαλλοντολόγοι του κάνουν το βίο αβίωτο. Επίσης, ε, η συγκέντρωση του διοξιδίου του άνθρακα ε, στο, στην καλλιέργεια βρίσκεται κυρίως ε, ε, στον Ισημερινό που δεσμεύεται πάνω από την Ισημερινό, στα τροπικά δάση. Αν θέλουμε λοιπόν να κάνουμε πραγματικά κάτι για τα αέρια του θερμοκηπίου, κάντε κάτι για τα τροπικά δάση. Εκείνη που υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα, όχι στι γεωργικέ φάρμε. Θα πρέπει να εκτιμούμε το διοξίδιο του άνθρακα, γιατί το χρειάζονται τα φυτά για την ε, τροφή τους. Δεν θα πρέπει να το κατηγορούμε έτσι. Ο κύριος Φλάναγκαν. Ακούμε διαρκώς, είτε είναι σωστό είτε όχι, ότι θα πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των γεών για κάθε εκτάριο να υπάρχει μέγιστη απόδοση εγώ από αυτά που έχω ακούσει τις τελευταίες εβδομάδες, αν θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό, το να φυτεύει κανείς δέντρα για την ε, παραγωγή ενέργειας ε, με καύση μετά των δέντρων από τη γη του καθενός, δεν είναι πιο αποτελεσματική χρήση των εκταρίων αυτών και είναι απλό. Αν αντί να ε, φυτεύουμε δέντρα και να τα καίμε μετά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη γη αυτή για φωτοβολταϊκά είναι επιστημονικό γεγονό ότι έτσι παράγεται πιο πολλή ενέργεια. Πώ το αμφισβητούμε αυτό, αλλά φαίνεται ότι η πολιτική αντίθεται στην παρούσα φάση σε αυτό. Πώ γίνεται λοιπόν αυτό η πολιτική, δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά σε μια νέα θρησκεία. Η θρησκεία είναι ότι έχω επενδύσει στην περιοχή αυτή και κάτι θα πρέπει να βγάλω. Ανεξάρτητα από το πόσο γελία θα είναι η λύση που θα επιλέξω και σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα. Πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά την περιοχή μου είχα προωθήσει τις ιδέες αυτές στην περιοχή μου και ήμουν βλάκας. Να επαναλάβω κάτι που είπε ένας οικονομολόγος στην Ιρλανδία για διαφορετικό θέμα. Αν ε, κανείς ε, με το αυτοκίνητο του μπει σε ένα χαντάκι, δεν συνεχίζει να πηγαίνει μπροστά. Κάνει βάση όπισθεν και προσπαθεί να βγει από το χαντάκι. Άρα πιο πολλή ενέργεια μπορεί να, παραχθεί από άλλες τεχνολογίες, από την πολύ βασική τεχνολογία της καύσης ξύλου. Θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε θρησκευτικοί στα πιστεύω μας και να εφαρμόσουμε επιστημονικές αρχές. Σε Το θέμα της ενέργειας συνδέεται στενά με το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Ε, στο εσωτερικό αυτό, με αυτό το, δεδομένο, τα κράτη-μέλη έχουν κάποιες ε, επιλογές ε, στον ενεργειακό αυτό Θα πρέπει μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση να μας επιτρέπει να δούμε το παγκόσμιο θέμα ενέργεια, κλιματική αλλαγή, που είναι αλληλένδετα οι επενδύσεις. Φυσικά χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το θέμα των βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς σε σχέση με τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς. Και τα βιοκαύσιμα της πρώτης γενιάς ε, χρειαζόταν πραγματικά πολλές επενδύσεις, ε, οι οποίες δεν έχουν αποσβεστεί ακόμα και η διάρκεια της ε, απόσβεσης είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουμε συμφέρον να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για τις επενδύσεις αυτές. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα. από την Αρμόδια Γενική Επιτροπή. Ο Διευθυντής, ο κ. Σπίρχοου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ονομάζονται Βάικμαν από την DG Κλίμα και θα μιλήσει και η συνάδελφος από την DG Έρευνας. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Μάλιστα, είναι κοινή πρόταση από τις δύο γενικές διευθύνσεις, λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ε, Σκοπό Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι αποτελεσματικός ο τρόπος επίτευξης των στόχων της Ενεργειακής Ένωση. Θα είναι σύντομο. γιατί το σχέδιο έκθεση ήταν και αυτό αρκετά σύντομο. Γνέρουμε, ξέρουμε ότι ο, μάλλον σημειώνουμε ότι ο εισηγητής ε, καλώς ορίζει την πρόταση ως ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και σκοπεύουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο από πλευρά τη Επιτροπή ε, προ την κατεύθυνση αυτή σε ό,τι αφορά το, το LULUCF, τη συγκεκριμένη πρόταση. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν οι προτάσει αυτέ και θα τι εξετάσουμε σε συνάρτηση και με τι υπόλοιπε προτάσει. Και είναι σημαντικό επίση να σημειώσουμε και το αίτημα για σταθερότητα το οποίο αναφέρθηκε στην τελευταία παρέμβαση είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την πρόταση αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει σταθερότητα για τους επενδυτές αν θέλουμε να προβαίνουν πραγματικά σε επενδύσεις για να κάνουμε και τη μετάβαση στην ε, οικονομία χαμηλής εκπομπής άνθρακα. Και σκοπός μας ε, δεν είναι να μεταφερθούν ε, Δραματικέ αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό τη μπορεί να πετύχει του στόχου τη ε, σε ό,τι αφορά το κλίμα και την ενέργεια. Η συνάδελφο θα ήθελε μήπως να πάρει το λόγο να προσθέσει κάτι. Ναι, σα ευχαριστώ, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο σα αγαπητή Επιτροπή και βλέπουμε πραγματικά ποιο είναι ο ρόλο τη Γεωργίας. Πολύ σημαντικό, σημαντικός κλάδος σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση τη Ενεργειακή Ένωση και αυτό αποτυπώνεται και στι προτάσει σα Να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή για τα σχόλιά του, τα οποία ήταν πολύ στοχευμένα. Συγκεκριμένα για την πρόταση να υπάρξουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και εκτάσεις για την βιοενέργεια. Το έχουμε λάβει υπόψη αυτό και υπάρχει και μία πρώτη αγραφή βάση μιας ε, Εκτελεστικέ πράξει και θα χρειαστεί να τα εξηγήσουμε αυτά με μεγαλύτερη σαφήνεια, αλλά τεχνικός πώ τι αναμένουμε από την υποβολή εκθέσεων αυτή σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε για τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα αντικαταστήσουν τι κατευθυντήριε γραμμέ και τι συστάσεις. Υποστηρίζουμε την τη φιλοδοξία, αυτό σίγουρα. Όσο και να θα θέλαμε, και αν θα θέλαμε να υπάρχει κάτι δεσμευτικού χαρακτήρα όταν αξιολογούμε στην πρόοδο των σχεδίων των κρατών μελών, αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο όπου συζητάμε ευρωπαϊκούς στόχους και δεν υποστηρίζεται αυτό από τους εθνικούς στόχους, το οποίο και περιπλέκει την κατάσταση. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, δεν προτείναμε κάτι τέτοιο στην αξιολόγησή μας ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη συμπερίληψη δεσμευτικού χαρακτήρα διαγραφών και λέμε ότι τα κρατημέρια θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις συστάσεις και φυσικά επιφυλασσόμεθα επιφυλάσσονται μάλλον τα κρατημέλη να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση που οι συστάσεις αυτές δεν λαμβάνουν αρκετά υπόψη στα σχέδια. Να τονίσω επίσης ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας σε ό,τι αφορά και τις ε, συστάσεις των, ευρωπαϊκών, των εθνικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων και των εθνικών ε, βουλών. Δεν ε, τέθηκαν θέματα επικουρικότητα σε ό,τι αφορά την διαχείριση, της διακυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τη δημόσια τώρα διαβούλευση. Αυτή θα καθοριστεί από τα κρατημέλη οι λεπτομέρειες αυτή θα καθοριστούν από τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη δουλειά σας και προσβλέπουμε στην ε, συνεργασία μαζί σας και περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σρόντε. Σας ευχαριστώ. Μια και έμεινα τελικά. Θα ήθελα να πω δύο λόγια. Προς τον κύριο Γιάρα και προς τους άλλους συναδέλφους θα ήθελα να τους εμπιστήσω την προσοχή στο εξή. Η έκθεση αυτή και αυτή η γνωμοδότηση πρόκειται και αφορά μόνο θέματα διακυβέρνησης ε, ή τα θέματα ουσίας. Περιλαμβάνονται με μεμονωμένες εκθέσεις και στις μεμονωμένες νομοθετικές προτάσεις. Αυτό, κυρίε και κύριοι, μιλάμε αμυγός για διακυβέρνηση, να το έχουμε αυτό υπόψη. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα μεμονωμένα ζητήματα. δεν θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε άλλωστε όλα αυτά στην εγγραμματοδότηση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θέματα διακυβέρνηση, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου προ αυτά που είπε ο κ. Δελκάστρο. Ότι ασφαλώ και χρειαζόμαστε το μέγιστο σε διαφάνεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε. Μέχρι 27 Ιουνίου στη μία το μεσημέρι μπορείτε να καταθέσετε τι τροπολογίε σα. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό. Το επόμενο το σημείο 9 έχει αναβληθεί. Οπότε θα διακόψουμε μέχρι τις 11.30 που θα συνεδριάσουν και κλεισμένο των θυρών οι συντονιστές. Η υπόλοιπη επιτροπή θα ξανασυνεδριάσει στις τρεις έχουμε σημαντική παρουσίαση έκθεση και μετά συνάντηση με δύο επιτρόπους. Ε, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συντονιστές, αν γίνεται, να μην περιμένουμε σε δεκάμιση αλλά να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα τη δική του συνεδρία. Ευχαριστώ. συγγνώμη, ο κύριος Άγνιο. Μία διευκρίνηση. Πότε θα ξεκινήσουν τελικά οι συντονιστές την δική του συνεδρίαση. Μπορείτε να μας το προσδιορίσετε. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος. Αν γίνεται 11 παρατέταρτο, 11 παρατέταρτο, αν συμφωνούν οι συντονιστές και ευκαιρούν, να ξεκινήσουμε 11 παρατέταρτο συνεδρία των συντονιστών. Ο κύριος Νίκολσον. Ναι, αλλά δεν θέλω να είμαι γεννής, αλλά έχουμε ε, προβλέψει άλλε συνεδριάσεις ενδιάμεσα. Θα προσπαθήσω, αλλά πρέπει να αλλάξω. Καλά, τότε 11. 11. 11 θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Μια και δεν συμφωνούμε για 11 παρατέταρτο, θα ξεκινήσουμε 11 η ώρα τη συνεδρίαση των συντονιστών.